η αναγνώριση από την Κροατία και την Κύπρο ορισμένων εγγράφων και ούτω κατεξής. Η κυρία Τάνια Φατζόν είναι η συγγήτρια. Και εδώ ψηφίζουμε επί του κειμένου. Α, όχι, βλέπω υπάρχουν κάποιες τροπολογίες. Για να δούμε τις τροπολογίες, παρακαλώ. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Τι Σχόλια εκτός μικροφώνου. Δεν ακούτε τα γαλλικά. Πώς γίνεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε επί της τροπολογίας Πέντε 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Λάθος μου. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτή τη φορά τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική λοιπόν ψηφορία, έναρξη ψηφορίας. Πέρας ψηφορίας. Ομοφόνος με 44 ψήφους υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Κυρία Φατζόν, συγχαρητήρια. Και εντολή διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Ξέρετε μια ψηφή υπέρ, 0 κατά μηδέν εποχές. Ομοφόνος επίσης. Κύριε Φατζόν, συγχαρητήρια και πάλι. Αυτά ως προς τις ψηφοφορίες. Now, we turn back. Και επανερχόμεθα στα δικά μας, σημείο 14. Έρευνα τη Επιτροπή σχετικά με την ηλεκτρονική μαζική επιτήρηση πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τι ρωσικέ μεθόδου υποκλοπή των επικοινωνιών. Έχουμε εδώ το κύριο πιάτο για σήμερα. Μαζικέ υποκλοπέ. παρακολούθηση πολιτών. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντρέη Σολντατόφ, ερευνητής επί ερευνητής δημοσιογράφος, ο οποίος ε, ειδικεύεται στο θέμα. Είναι μαζί μας ε, από τη Μόσχα, μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρακαλώ ησυχία, ώστε να φύγουν με ησυχία. Παρακαλώ για να ακούσουμε τον κύριο Σολντατόφ από τη Μόσχα. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ε, τηλεδιάσκεψη. Όσοι θέλουν να φύγουν, επαναλαμβάνω, όσο πιο ήσυχα γίνεται. Κύριε Σολντατόφ, με ακούτε? Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Χαιρετούμε τη Μόσχα. Αν είστε έτοιμος, σας ακούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω να βλέπετε τις διαφάνειες. Πού είναι οι διαφάνειες, λέει πρόεδρος. Δεν, δεν, δεν τις βλέπω εγώ τουλάχιστον. Πρόεδρος, για να δούμε εάν έχουμε σύνδεση. Πολύ ωραία, όχι, βλέπουμε τις διαφανίες σας. Ωραία, εξαιρετικά. Προχωρήστε. Τεχνικές παρακολουθήσεις της Ρωσίας. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Να συστηθώ καταρχήν. και γιατί ασχολούμαι με τις πρακτικές παρακολούθησης. Είμαι ερευνητής δημοσιογράφος με βάση τη Μόσχα, υπευθύνω για τον ιστορικό agentura.ru. Παρακολουθούμε τις ε, ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Δημιουργήσαμε το δίκτυό μας το 2000. Ξεκινήσαμε από το Λονδίνο. Uh, surveillance. Uh, the next slide, please.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 Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αντικατασκοπίας, η κυρία Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και η ORM είναι η τεχνική ομάδα η οποία κάνει τις παρακολουθήσεις. Το σύστημα SORM είναι ένας ε, ρωσικός φορέας που κληρονομήσαμε από τη Σοβιετική Ένωση χρονολογείται από, τα, από τη δεκαετία του 80. Φυσικά έχει προσαρμοστεί στις ε, νέες ανάγκες και νέες τεχνολογίες. Στο διαδίκτυο, στην παρακολούθηση του Skype, των κινητών τηλεφώνων, τα δίκτυα τρίτης γενεάς και ούτω καθεξής. Πρόκειται όμως για που επαναλαμβάνω της Σοβιετικής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα γεννήθηκε μέσα σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Αυτό εξηγεί και ορισμένα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα, όπως για παράδειγμα τα σχετικά εντάλματα παρακολούθησης. Τα στελέχη της FSB χρειάζονται βεβαίως ένταλμα για να προβούν σε παρακολουθήσεις. Το πρόβλημα είναι όμως ότι τα στελέχη της FSB δεν είναι υποχρεωμένα καν να επιδείξουν το σχετικό ένδελμα και ιδιαίτερα στους παρόχους τηλεπικοινωνικών υπηρεσιών. Υποχρεούνται να το επιδείξουν στο δικαστήριο, αλλά όχι σε κανέναν άλλον. Οι πάροχοι και οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών υποχρεούνται να πληρώσουν για το κόστος του ΣΟΡΜ. Δεν έχουν όμως την ε, δυνατότητα να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του ΣΟΡΜ. Η FSB είναι συνδεμένη σε κάθε πόλη με ειδικά καλώδια με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην περιοχή. Από τεχνολογικής απόψεως λοιπόν, η κατάσταση είχε εξή. Υπάρχει διαφορά στην τεχνική προσέγγιση μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Στην Ευρώπη, όπως βλέπετε εδώ, έχετε δύο γραμμές επικοινωνίας μεταξύ της αστυνομία για παράδειγμα και των παρόχων. Επάνω βλέπετε την εντολή προς τον πάροχο τηλεπικοινωνικών υπηρεσιών που παρακολουθεί και μέσω μιας δεύτερης γραμμής αποστέλει τα δεδομένα στην αστυνομία. Στη Ρωσία οι νόμιμες παρακολουθήσεις γίνονται μέσω ενός καναλιού και μόνο. Βλέπετε ότι συνδέεται ο πάροχος με τα γραφεία του FSB. Τεχνικός, το στέλεχος του FSB μπορεί να ξεκινήσει μια παρακολούθηση με δική του πρωτοβουλία να σταματήσει την παρακολούθηση, να προσθέσει ονόματα, για παράδειγμα, χωρίς να λάβει γνώση ο πάροχος τηλεπικοινωνικών υπηρεσιών. Έτσι ο πάροχος δεν γνωρίζει ποιος παρακολουθείται και πότε. Και τούτο, χάρη στο γεγονός ότι η FSB έχει εκ του μακρόθεν δυνατότητα παρακολούθησης με απευθείας παρεμβολή στους κεντρικούς υπολογιστέ του παρόχου. Ποιοι είναι οι χρήστες του SORM. Βάσει νόμου, 8 υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν παρακολουθήσεις το Υπουργείο Εσωτερικών, η FSP, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας, η Υπηρεσία Αντικατασκοπίας, τα Τελωνία, η Υπηρεσία Κρατών Ναρκωτικών, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών και η Αντικατασκοπία του Γενικού Επιτελείου. Από τη δεκαετία του 90 πάντως αποφασίστηκε από τον Γέλσιν και την κυβέρνησή του η FSB να διαχειρίζεται το σύστημα SORM. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν οι άλλες υπηρεσίε πρέπει να παρακολουθήσουν κάποιες επικοινωνίες, πρέπει να επικοινωνήσουν με την FSB και έτσι να οργανωθεί η παρακολούθηση συγκεκριμένου, για παράδειγμα, προσώπου. Η FSB, λοιπόν, από τεχνικής απόψεως, διεξάγει την παρακολούθηση. Αυτά Τη δεκαετία του 90 και του 2000. Τα πράγματα εν συνεχεία άλλαξαν. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι καταρχήν η σημαντική αύξηση των παρακολουθήσεων τηλεφώνων και email. Βλέπετε εδώ τα επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα τελευταία 6 χρόνια το πλήθος των παρακολουθήσεων διπλασιάστηκε. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτές τις στατιστικές δεν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες αντικατασκοπίας. Δεν περιλαμβάνονται λοιπόν οι ξένοι, οι δημοσιογράφοι και άλλοι. Η πρώτη ενημέρωση, η αναβάθμιση του συστήματος έγινε διαφορετικά ως εξή. Όπως ε, προείπα, η FSB δίκη το SORM. Η κατάσταση όμως αυτή άλλαξε στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Όταν αναλύσαμε τις συμβάσεις που είχε υπογράψει η κυβέρνηση, διαπιστώσαμε ότι τρεις άλλες υπηρεσίες είχαν αρχίσει να δημιουργούν τα δικά τους αντίστοιχα SORM. Οι τρεις αυτές υπηρεσίες είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, η Υπηρεσία κατά των Ναρκωτικών και η Υπηρεσία των Φυλακών. Επόμενη διαφάνεια. Ένα από τα ερωτήματα είναι, είναι κατά πόσον το ΣΟΡΜ χρησιμοποιείται κατά τη αντιπολίτευση. Κάθε φορά που έβγαινε ε, κάτι στις ρωσικές εφημερίδες, ε, η κυβέρνηση έλεγε ότι εμπλέκονται δημοσιογράφοι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης παρακολουθήθηκε από το ΣΟΡΜ να μην σας διαβάζω τώρα όλα αυτά τα παραδείγματα, αλλά το ανώτερο δικαστήριο και όχι μόνο τα τοπικά δικαστήρια ενέκριναν την απόφαση της FSB να παρακολουθεί ακριβώς τις επικοινωνίες συγκεκριμένου βουλευτή ο οποίος παρακολουθεί το μόνο και μόνο επειδή είχε λάβει μέρος σε συλλαλητήριο το οποίο ήταν επικριτικό κατά της FSB. Την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ελπίζω να με ακούτε. Το θέμα στις μέρες μας βεβαίω, το μεγάλο θέμα είναι το σόκι. Τα σχετικά δημοσιεύθηκαν στην Guardian τον Οκτώβριο, σχετικά με το σύστημα δηλαδή, το οποίο εγκαταστάθηκε στο Σότσι εν Ολυμπιακών. Δεν είναι μόνο οι κάμερες, τα κλειστά κυκλώματα και άλλα μέτρα αλλά το ίδιο το ΣΟΡΜ. Το 2010, όπως είπα, η FSB ετέθη επικεφαλής της ασφάλειας των Ολυμπιακών και ζητήθηκε το ΣΟΡΜ να αναβαθμιστεί ειδικά για να ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες των επισκεπτών του Σότσι. Διαπιστώσαμε ότι υπηρεσίες όπως η Roscom Nasdor επαλήθευσαν τη λειτουργία του εξοπλισμού της SORM για να δουν αν τα συστήματα λειτουργούν ικανοποιητικά εν ώψη των Ολυμπιακών. Ένα τελευταίο σχόλιο. Το SORM δεν είναι μόνο ρωσικό πρόβλημα και θα εξηγήσω γιατί. Ακόμη και σήμερα η νομοθεσία περί μυστικών υπηρεσιών χρονολογείται από τη Σοβιετική Ένωση. και αφορά και πρώην χώρε τη Σοβιετική Ένωση, ειδικά όσον αφορά τι υπηρεσίε αντικατασκοπία. Το ΣΟΡΜ φαίνεται ότι χρησιμοποιείται και σε αυτέ τι χώρε. Τοπικά δηλαδή ΣΟΡΜ χρησιμοποιούνται στην Λευκορωσία, την Ουκρανία, το Ουσμπεκιστάν, το Κυριστάν και το Καζακστάν. Επόμενη διαφάνεια. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σολδατόφ. Για τι απόψεις σας, ως συνήθως, ερωτήσεις, απαντήσεις. Ας δούμε λοιπόν ποιοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Σηκώστε τα χέρια παρακαλώ. Μωράς. Όχι. Διαδικαστικό πρόεδρε. Δεν είχαμε διερμηνία της ομιλίας αυτής. Σε καμία γλώσσα. Ούτε οι άλλοι τα άκουσαν. Σε καμία γλώσσα δεν βγήκε η διερμηνία. Ζητώ συγγνώμη. Λυπάμαι. Μόνο αγγλικά ακουγόταν. Δεν υπήρξε, λέει, ο πρόεδρος ε, μετάφραση σε καμία γλώσσα. Όλες οι καμπίνες δούλευαν, πάντως η ελληνική καμπίνα δούλευε. Δεν ξέρω ίσως αν υπήρχε πρόβλημα με κάποιους ευρωβουλευτές, οι οποίοι δεν έβαλαν τα ακουστικά τους. Θα μιλήσει ο κ. Μωρές, ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους γιατί γίνεται αυτή η συνέντευξη για το θέμα των παρακολουθήσεων από τη Ρωσία ε, λόγω των ανησυχών που έχουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι και πιθανών δραστηριοτήτων και για πιθανές δραστηριότητες της FSB αλλά και, και άλλων υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Η ερώτησή μου αφορά την παρακολούθηση στο Σότσι όπως αναφέρεται από τον Guardian ότι έχει οργανωθεί, αλλά επίσης θέλω να ρωτήσω πόσο εκτεταμένο μπορεί να είναι το φαινόμενο αυτό σε σχέση με ευρωπαϊκές παρακολουθήσεις. Δεν επεκταθήκατε τόσο πολύ στο θέμα των σοβιετικών ε, δορυφόρων. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο βαθμό ή πόσο πέραν των δορυφόρων υπάρχει. Κοιτάξτε, το σόρμα χρησιμοποιείται κυρίως στο ιστορικό μιας χώρας. Της χώρας δεν είναι ένα σύστημα παρακολούθησης στο εξωτερικό. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ε, χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα για την παρακολούθηση εκτός Ρωσίας, αλλά ασφαλώς μπορούν να το αξιοποιήσουν το σόρμ για τις χώρες. Διότι όταν αποφασίσουν. Όταν αποφάσισαν να βγουν από το σύστημα αυτό το σοβιετικό και να προσεγγίσουν ε, τα συστήματα παρακολούθησης, ε, λήφθησαν αποφάσεις. Μπορεί οι ρωσικές εταιρείες να ήταν αυτές οι οποίες προσέφεραν τις καλύτερες επιλογές για την εσωτερική παρακολούθηση των χωρών αυτών, γιατί γνωρίζουμε ότι του τους τρόπους ε, των, ε, του εξοπλισμού σόρμα. Άρα μπορεί να γνωρίζουμε καλύτερα από τι ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές χώρες ε, τι είδους συστήματα χρειάζεται, το Ουσβεκιστάν, το Καζακστάν, η Ουκρανία κτλ. Αλλά πάντως το ΣΟΡΜ περιορίζεται στην επικράτεια της πρώην Σοβιετικής Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόλτατοφ. Η τεχνική υπηρεσία η οποία αναλαμβάνει τεχνική υποστήριξη της ε, ε, διερεύνηση αυτή για τις μαζικές παρακολουθήσεις της Επιτροπής μας μας επισημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα τεχνικό για ε, στην διερμηνία και άρα δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον ήχο αυτή της παρουσίαση με τι διαφάνειε, Λέει ο πρόεδρος, οι διερμηνεί το παρακολουθούσαν. Πρέπει να πούμε Εν πάση περιπτώσει υπάρχει δυσκολία ως προς την παρακολούθηση της διερμηνίας της γλώσσας. Εάν κάτι μπορεί να κάνει τεχνική υπηρεσία, παρακαλούμε να αναλάβει τις σχετικές, τα σχετικά μέτρα για να παρακολουθούμε όλοι. Εγώ προτείνω, κύριε Σόλδατοφ να λάβετε, να σημειώσετε τις ερωτήσεις που θα διατυπώσουν οι σκιώδεις ηγητές. Να σημειώσετε τις ερωτήσεις λοιπόν και μετά θα δώσω το λόγο σε εσά για να πατήσετε σε όλες τις ερωτήσεις μαζί, αν συμφωνείτε. Ο κύριος Φως, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις, όχι πολύ Εάν συγκριθούν οι δραστηριότητες της NSA με αυτές ε, τις, ε, τις υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών της χώρας σας, πώς θα τις βλέπατε, τι είδους διαφορές εντοπίζατε. Δεύτερον, μετά τις επιθέσεις στο Βόλκοκρατ, η κοινή γνώμη στη Ρωσία, τι στάση τηρεί, εάν τηρεί. Και τρίτον, υπάρχει κάποιο σύστημα ισοδύναμο με αυτό της παρακολούθησης της επιχειρήσεις βιομηχανική κατασκοπία της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Φως και για τις προσπάθειές σας να μιλήσετε στα αγγλικά. Εγώ αυτό προτείνω όσο δεν έχει λυθεί το τεχνικό πρόβλημα. Επαραλαμβάνει ο πρόεδρος ότι οι διερμηνείς δεν είχαν αρκετό επίπεδο, αρκετή, αρκετή ένταση ήχου στις καμπίνες. Μιλάμε αγγλικά λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, ε, γιατί ακόμη δεν μπορούν να παρακολουθήσουν διερμηνείς. Μάλλον υπάρχει κάποια παρεξήγηση, διερμηνείς παρακολουθούν πολύ καλά. Κυρία Νετφέλτ, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Σολτατόφ που ήρθατε να μα μιλήσετε, που μα μιλάτε μάλλον σε αποστάσεω. Ε, σήμερα πρώτη μου ερώτηση λοιπόν. Σε σχετισμό με το Σότσι, τον οποίο σχετισμό ήδη αναφέρατε εσείς και είπατε ότι υπάρχει αυτή η ενίσχυση της εξωτερικής παρακολούθησης, αλλά πέραν της, αλλά μπορούμε να το διαχωρίσουμε αυτό από την εξωτερική παρακολούθηση. Και μήπως υπάρξει ο πειρασμός άπαξ εγκατασταθεί το σύστημα και αξιοποιηθεί στην περίπτωση του Σότσι, να επεκταθεί το πρόγραμμα. Έχετε την καλοσύνη, είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε. Μήπως επεκταθεί λοιπόν και για παρακολούθηση εκτός. Έχετε κάποια γνώση κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συστήματα μαζικής παρακολούθησης, την αυτά το SORM ή κάτι άλλο. Έχετε λοιπόν υπόψη πρόσβαση ενδεχομένω από πλευρά των ρωσικών αρχών για μαζική παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών των των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, βλέπετε να υπάρχει κάποια δυνατότητα εποπτείας σε παρακολούθηση ελέγχου από κοινοβούλιο που να έχει βέβαια κάποιο αποτέλεσμα. Και επίσης υπάρχει κάποια δυνατότητα από το Συμβούλιο της Ευρώπης όπου παραμένει μέλος η Ρωσία και για το οποίο θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ κύριε Ντφέλτ. Ο κύριος Άλμπρεχτ δεν είναι εδώ. Είχε άλλες υποχρεώσεις ενελειμμένες. Θέλει κανείς το λόγο για εκ μέρους των Πρασίνων. Όχι. Ο κύριος Κίρκοπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Σολτατόφ. Ευχαριστώ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Ασφαλώς όλοι μας εδώ ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους Ολυμπιακούς της Ότσι. Και κάποιοι από εμά επίσης αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει όντως ανάγκη οι αρχές της Ρωσίας να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία αυτών που συμμετέχουν στους αγώνες. Έτσι λοιπόν και με δεδομένα τόσα μας είπατε, ασφαλώς και θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποια δομή βάσει τη οποία θα εξασφαλίζουν αυτή την προστασία, θα συμμετέχουν σε αυτή, στο χώρο προστασία οι μυστικέ υπηρεσίε. Ε, Πάντω, μια και μα μιλάτε από καρδία σήμερα, δεν θέλω να ρωτήσω το εξή. Έχετε υπόψη σας πώς αντιδρούν στη σημερινή σας ε, τοποθέτηση σήμερα οι αρχές και εσείς ως ερευνητής δημοσιογράφος έχετε επαφές έμεσες ή άμεσες με τον κύριο Έντουαρτ Σνόντεν, ο οποίος από ό,τι γνωρίζουμε βρίσκεται στη Ρωσία. Έχετε συζητήσει μαζί του, σας έχουν επιτρέψει οι αρχές το ερευνητικό σας έργο, στα πλαίσια του ερευνητικού σας έργου, να συζητήσετε μαζί του ε, ενδεχομένες ανησυχίες που έχει για την ηλεκτρονική παρακολούθηση και τη θέση της NSA. Και βεβαίως θα θέλω να πω ότι αντιλαμβάνω πως μιλάτε ελεύθερα και από καρδία σήμερα. Ε, μπορείτε να μας κάνετε μια συγκριτική ανάλυση της δομής, ιστορικής δομής της ε, ΚΑΓΕΜΠΕ και της τωρινής πιο ελεγχόμενης δομής της FSB, ε, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας. Από τώρα. Ernst, κυρία Ernst. Δεν είναι εδώ όμως. Ε, τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Σολτατόφ και συνεχεία θα ξαναδώσω το λόγο στου ευρωβουλευτέ για περαιτέρω ερωτήσει. Uh, let's start with the first question, uh, comparison uh, between NSA activity and the FSB activity. I think that um, given the revelations made by Mr. Snowden, especially about the prison program, it seemed to me uh, that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 like border troops and electronic intelligence service, and it's the most mighty and powerful security service in the country. Well, I think that's all. Thank you, Mr. Soldatov. Ευχαριστώ κύριε Σολτατόφ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για να τεθούν και άλλες ερωτήσεις από ευρωβουλευτές. Θα συμμετάσχουν λοιπόν και άλλοι ευρωβουλευτέ στην συζήτηση. Η κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το δημοσιογράφο τι απαντάει στα νέα που βγήκαν για τις απειλές που έχει δεχτεί ο Έντουαρτ Σνόντεν. Πιστεύετε ότι αυτά τα νέα, αυτές οι ειδήσει είναι αξιόπιστες. Εσείς τι ξέρετε γι' αυτό. Υπάρχει κίνδυνο για το Σνόντεν, ο οποίος όπως λέτε είναι προστατευόμενος. Έχετε λοιπόν κάποιες πληροφορίες για αυτά τα νέα, για αυτές τις ειδήσει που, προέκυψαν. Κύριε, Σολτα... Κύριε Σολτατόφ, σας ε, μετέφρασαν την ερώτηση της κυρίας ε, Ρομέρο Λόπεθ. Θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. κυρία Γκόμες, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Σολτατόφ, είπατε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα, καλύτερα, η FSB, η Ρωσική, να κατασκοπεύσει, να παρακολουθήσει μαζικά την Ευρώπη. Ξέρετε αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για να ε, κατασκοπευθούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ας πούμε έκανε η Αμερική με την κυρία Μέρκελ. Χθε επίσης ακούσαμε στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, εξωτερικών υποθέσεων δηλαδή, ότι κάποιοι διαδηλωτές στο Κίεβο της Ουκρανίας, σε μια κεντρική πλατεία του Κιέβου, έλαβαν μηνύματα από τις αρχές που τους ε, έλεγαν «Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι είστε εδώ, είστε υπόλογοι». Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να περάσει αυτό το μήνυμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους, στους ανθρώπους που επιθυμούν οι αρχές. Είναι δηλαδή αυτός ο τρόπος επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι Ουκρανικές αρχές ρωσική τεχνολογία. Επίσης, τώρα δεν υπάρχει ο έλεγχος ε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ε, όπως ας πούμε υπήρχε με την ΚΑΓΕΜΠΕ, τώρα προφανώς η FSB δεν ελέγχεται από κάποιο κόμμα. Υπάρχει κάποιος ε, κοινοβουλευτικός έλεγχος από την Ρωσική Ντούμα της FSB. Θέλει κάποιος άλλος να υποβάλει ερώτηση. Η κυρία Ιντβελτ, ξανά. Αφού έχουμε χρόνο, να κάνω και άλλες ερωτήσεις. Είπατε ότι η NSA έχει κάποιο φυσικό πλεονέκτημα. Γιατί σε, πολλούς, σε πολλές χώρες ε, το αμερικανικό λογισμικό και οι αμερικανικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται, όποια και αν είναι αυτή η χώρα. Φαντάζομαι ότι και στη Ρωσία όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται αμερικανικά προϊόντα. Αυτό διευκολύνει τη σύνδεση με συστήματα που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη τότε και σε άλλες χώρες του κόσμου. Και κατά την άποψή σας, αυτό επιτρέπει στην FSB να επεκτείνει τις δραστηριότητες παρακολούθησης εκτός της Ρωσίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη ερώτηση. Με έκπληξη άκουσα να λέτε ότι όχι μόνο θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα για να υποκλαπούν επικοινωνίες, στο Σότσι και γύρω από το Σότσι, αλλά και τα μέτα δεδομένα τα οποία θα συλλεγούν θα αποθηκευτούν για τρία χρόνια. Από ό,τι ξέρετε, οι συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς, κυρίως για τις ευρωπαϊκές χώρες με ενδιαφέρουν, ε, Κάποιοι από τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκές έχουν γύρει κάποιες αντιρρήσεις σε αυτό. Φαντάζομαι ότι θα είναι ενημερωμένες. Είπε κάποιος κάτι, κάποιος υπουργό Εξωτερικών, Ήρθε σε επαφή με τη ρωσική κυβέρνηση να διαμαρτυρηθεί γι' αυτό, να γύρει οποιαδήποτε αντίρρηση. Σας κάλυψα όλους, πήρατε όλοι το λόγο. Αν ναι, ο κύριος Σολτατόφ μπορεί τώρα να απαντήσει στις τελικές ερωτήσεις πριν δώσουμε ξανά το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. First, uh, about Snowden and, uh, and, and threats. Uh, I don't think that these threats are genuine just because, uh, well,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 για τη συμμετάσχεση, το χρόνο σας να συμμετάσχετε σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Κύριος Μωρές, έχετε κάποια παρατήρηση? Όχι. Τώρα φτάσαμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χαιρετούμε. Εκτιμώ πολύ την αξία των παρατηρήσεών σας. Ευχαριστώ. Προχωρούμε. Επόμενο σημείο. Στην ημερήσια διάταξη δεν έχουμε έρευνες πλέον, αλλά απαλλαγή προπλησμός του 2012. Έχουμε εδώ αριθμό εκθέσεων. Η κυρία Ρότοβα η οποία είναι εδώ μαζί μας σήμερα και η κυρία Ματιό είναι συνεισηγητρίας. Και είναι η συζήτηση λοιπόν για επόμενα 40 λεπτά. Απαλλαγή των τομέα βεβαίω δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων και για την Eurojustin Frontex, το Ευρωπαϊκό Κολέγιο, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, το European Police Office, την Europol δηλαδή κλπ. Και την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Επιτήρησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έχουμε εδώ διάφορες υπηρεσίες, το Κέντρο Εποπτείας για τα Ναρκωτικά, καθώς και το Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Λοιπόν, να ακούσουμε τις ε, συνεισηγήτριες και μετά να συζητήσουμε. Κύριε Ρότοβα, καταρχήν, παρακαλώ. Πρόεδρε, σχέδιο γνωμοδότησης απαλλαγής για τον προπολογισμό των ε, σχετικών οργάνων θα ήθελα να υποβάλω τα τρία έγγραφα για μια κοινή συζήτηση. Γνωρίζω τις σχετικές υπηρεσίες και τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές δηλώνεται ότι οι λογαριασμοί των τριών υπηρεσιών αντικατοπτρίζουν πιστά τις ε, δημοσιονομικές υποχρεώσεις και ότι δεν υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις. Το ποσοστό σφάλματος είναι 4,8% όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του εκ ελέγχου. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί πηγή των λαθών. Εντοπίστηκαν όμως τα εξή ζητήματα στην Γενική Διεύθυνση HOME. Εντοπίστηκαν αποκλήσεις όσον αφορά το SIS, οι οποίες δεν ενεγράφησαν εντός της προθεσμίας. Το ίδιο ισχύει και το SIS 2 για διάφορους λόγους. Από την άλλη πλευρά σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη του SIS 2 του συστήματος πληροφοριών Schengen 2 δηλαδή. Η δεύτερη εκθέση αφορά την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εδώ εντοπίστηκαν δύο παραλήψεις, δύο προβλήματα. Η εκ των υστέρων επαλήθευση των δαπανών έγινε μόνο στο τέλος του 2012. Δεύτερον, η υπηρεσία. έχασε μια υπηρεσία, μια υπόθεση με συγχωρείτε ενώπιν του δικαστηρίου και πρέπει να βελτιώσει το χειρισμό των θεμάτων προσωπικού. Στην τρίτη έκθεση, όσον αφορά το κέντρο παρακολούθησης για τα ναρκωτικά, διαπιστώθηκαν πιο σημαντικά προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει ότι στο προ RADO δεν τηρήθηκαν οι κανόνες. Προσωπικά εκπλήτωμε διότι δεν έγιναν καθόλου έλεγχοι μετά το 2008, εκ των υστέρων έλεγχοι. Το πρόβλημα αφορά 200.000 ευρώ για χώρο που δεν χρησιμοποιείται στα παλιά γραφεία του οργανισμού. Αυτό είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα Θεωρώ ότι το κέντρο πρέπει να λύσει κατεπηγόντως το πρόβλημα αυτό. Τέλος, σημειώνω ότι το κέντρο δεν εφαρμόζει την ισότιμη εκπροσώπηση των υπαλλήλων από γεωγραφική Η Ιδιαίτερα δεν εκπροσωπούνται τα νέα κρατημέλη. Όλα αυτά περιγράφονται στην έκθεσή μου, όμως δεν ε, τροποποιούν την γενική άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου. Προτείνω λοιπόν την απαλλαγή. Θέλω να σα ενημερώσω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 27η Ιανουαρίου. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Χαιρετόφα, πολύ ωραία κυρία Μαρτιό. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε, όσον αφορά τις άλλες υπηρεσίες αρμοδιότητες της ΛΥΜΠΕ, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την Frontex για το 2012. Εδώ έχουμε κάποιες δυσκολίες. Το δικαστήριο δεν επιβεβαίωσε την νομιμότητα όλων των δραστηριοτήτων της Frontex. Και τούτο διότι η Frontex δεν υπέβαλε τα σχετικά δικαιολογητικά για την επαλήθευση των δαπανών σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Το ελληνικό συνέδριο σημειώνεται σχετικά Πρόκειται για συμβάσεις με εθνικές αρχές για τις αποστολές που υλοποιούν και που απαιτούν εξοπλισμό όπως ε, σκάφη θαλάσσης, αεροσκάφη κ.ο.κ. Η Frontex θεωρεί ότι η δήλωση των εθνικών αρχών αρκεί. Παρ' όλα αυτά, βάσει της κοινωτικής νομοθεσία, ο διευθυντής της Frontex είπε ήδη ότι για τις ε, περιπολίες για παράδειγμα θα θεσπίσει μια ωριαία χρέωση. Αυτό για το μέλλον. Δεν πιστεύω ότι αυτό πρέπει να επηρεάσει τη θετική μας άποψη για την απαλλαγή για το 2012. Για την Europol. Η Europol βελτίωσε σαφέστατα την ε, αναφορά ως προς τα χρηματοοικονομικά της. Μεταφέρθηκαν 7% ε, λιγότερα κονδύλια Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τον Ιούνιο του 2012 δημιουργήθηκε το Κέντρο Παρακολούθησης ε, του Κυβερνοχώρου. Η υπηρεσία βεβαίω προσαρμόστηκε στη νέα κατάσταση και προβλέπει ένα μέρος του προπολογισμού της για την αυτή υπηρεσία. Θα απαιτηθούν επιπλέον δραστηριότητες για να ολοκληρωθεί η απαλλαγή του 2011 και βεβαίω η υπηρεσία η Europol ε, είναι στη διαδικασία βελτίωσης των λογιστικών της για το ΣΕΠΟΛ υπάρχουν κάποια προβλήματα προπολογισμού και μεταφοράς πιστώσεων. Υπάρχει μια αβεβαιότητα προς το μέλλον της υπηρεσίας και ως προς το προσωπικό. Διευκρίνιζω επίσης ότι στην τροπολογία 5 υπάρχει ένα λάθος. Με την ευκαιρία όταν έρθει η ώρα θα υποβαλώ προφορική τροπολογία. Υποτίθεται ότι η ΣΕΠΟΛ θα συγχωνευτεί με την Europol. Αυτό δεν συνέβη ποτέ όμως. Περιμένουμε το ελληνικό συνέδριο, το Συμβούλιο με συγχωρείτε, να πάρει σχετική απόφαση, ώστε και στη συνέχεια η Κομισιόν να προβεί στη σχετική απόφαση. Περιμένουμε την απόφαση λοιπόν της Κομισιόν για να δούμε τι θα γίνει με τις εγκαταστάσεις ε, της ε, σε πόλη. Ελπίζω ότι η Κομισιόν να έχει απάντηση, μια που είναι παρούσα εδώ, να την ακούσουμε. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξη Ασύλου, εδώ έχουμε καθυστερήσει όσον αφορά την αναφορά των λογιστικών. Το 2012 η υπηρεσία έγινε ανεξάρτητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι είμαστε σε διαδικασία προσαρμογή λόγω τη πρώτη χρονιά αυτονομία, αν θέλετε. Επίση, η υπηρεσία προστασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι ακριβώ ανεξάρτητη υπηρεσία. Είναι μάλλον ανεξάρτητη ελεγκτική υπηρεσία. Εδώ δεν διαπιστώθηκε κανένα λάθο από το ελεγκτικό συνέδριο. Όσον αφορά τι αποζημιώσει, πάντω πρέπει να γίνουν μερικέ μικροβελτιώσει. Eurojust, όπω και πέρσι, Ζητούμε περισσότερη διαφάνεια στις διαδικασίες προσλήψεων. Ελπίζουμε ότι ήδη έχει μπει σε καλό δρόμο το θέμα. Τέλος, ζητούμε προσπάθεια, μια επιπλέον προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες για μια καλύτερη παρακολούθηση των διαδικασιών, περισσότερη πολυγλωσία για να μπορούμε να διαβάζουμε τα σχετικά στοιχεία και σε άλλες γλώσσες, όπως ε, εγώ. Προτείνω πάντως την απαλλαγή για τον σχετικό προπολισμό για όλες τις υπηρεσίες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τη θετική άποψη όσον αφορά την απαλλαγή για τους προπολογισμούς του 2012. Θέσατε μια ερώτηση όμως στην Κομισιόν. Να δώσουμε για δύο λεπτά το λόγο στην Κομισιόν για να την ακούσουμε πριν κλείσουμε τη σχετική συζήτηση. Κομισιόν μήπως θα ήθελε το λόγο. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ζητήματα που αφορούν την απαλλαγή προϋπολογισμού για την ε, Επιτροπή στους τομείς των εσωτερικών και της δικαιοσύνης. Άκουσα τις ε, παρατηρήσεις ε, ότι δεν δόθηκαν επαρκείς πληροφορίες εκτός από τον τομέα της δικαιοσύνης και εμείς συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά από την άλλη το ελεγκτικό συνέδριο οργανωτικά είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσδιορίσει τον ελεκτικό του δείγμα όπως καλύτερα μπορεί και εμείς βεβαίως μπορούμε όσο και αν θέλαμε να καλύπτουμε ολόκληρο τον προπολογισμό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Πάντως έχουμε τη λεπτομέρεια του δείγματο που χρησιμοποιήθηκε. Έγιναν εννέα επιλογές για τα εσωτερικά και πέντε για τη δικαιοσύνη και υπήρξαν κάποιες μικρές παρατηρήσεις που θεωρήθηκαν όχι αρκετά σημαντικές ώστε να περιληφθούν στην έκθεση. Ε, με ικανοποίηση σήμερα δεν υπάρχει παρατήρηση ως προς τη Γενική Διεύθυνση για τη Δικαιοσύνη, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει και το γεγονός ότι δεν είχαμε παρατηρήσει, δεν είχαμε προβλήματα στην έκθεση αυτή για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει πιο περίπλοκες, πιο περίπλοκες δομές και ευρεία λειτουργία και αρμοδιότητες για να απαντήσουμε στις συστάσεις της ε, του εσωτερικού ελέγχου που αφορούσε το μέσον Σέγγεν καθυστερήσαμε διότι δεν έγινε η... δεν έγινε αντιληπτή η θέση σε λειτουργία ε, της, ε, του μηχανισμού που αφορούσε την Κροατία από τους ελεγκτές. Γι' αυτό υπήρξε καθυστέρηση. Δηλαδή δεν ήταν σωστή τα ε, οι προθεσμίες, τα χρονοδιαγράμματα για τον εσωτερικό έλεγχο. Η έκθεση δραστηριοτήτων του 2012 ήταν τελευταία για την οποία εκφράζει επιφυλάξεις η Γενική Διεύθυνση ε, Εσωτερικών Υποθέσεων του 2013 όπως όλοι γνωρίζουν θα είναι πολύ πιο θετική και περιμένουμε ότι για το 2013 θα μπορέσουμε να εκφράσουμε ικανοποίηση και να άρουμε τις επιφυλάξεις μας για τους ε, λογαριασμούς. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος, για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μας δίνετε στα τόσο συναρπαστικά αυτά θέματα. Η κυρία Ματιού θα ήθελε να κάνει μια παρατήρηση, έχετε το λόγο. Ε, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ γιατί δεν έλαβα απόφαση, δεν απάντησε στην ερώτησή μου. Ενώ ακούσαμε απεγνωσμένες προτάσεις Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση, για την έδρα, την αλλαγή κυρίως έδρα του ΣΕΠΟΛ από πλευρά της Επιτροπής, τελικά δεν έγινε τίποτα. Και έπρεπε να φτάσουμε να περιμένουμε την απόφαση Πρόταση προς το Κοινοβούλιο από πλευράς του Συμβουλίου για την αλλαγή της έδρα για να, προχωρήσει η Επιτροπή και έτσι να κηρύξει έναν πόλεμο μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, Συμβουλίου και Επιτροπής, ατυχέστατο, που φέρνει και το Κοινοβούλιο σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό θέλω να μου δώσετε απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Σας ευχαριστώ, κυρία Ματσιό, για άλλη μια φορά. Έκανε μια πολύ σημαντική παρατήρηση κυρία Ματσιέ. Επιμένει και παρακαλώ την Επιτροπή να απαντήσει. Ναι βεβαίω. Ε, δεν ήμουν εγώ αρμόδια για την ερώτηση αυτή και γι' αυτό και δεν απάντησα. Έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις ως απάντηση. Είναι κάπως περίπλοκο το ζήτημα. Θα σας πρότεινα, και καταλαβαίνω βεβαίως ότι δεν είναι απλή κατάσταση, από πλευράς μας, Υπήρχαν σοβαροί λόγοι για τους οποίους χρειάστηκε να καθυστερήσουμε. Γιατί στόχος της Επιτροπής από τις πληροφορίες τουλάχιστον που έχω ήταν ανέκαθεν να εξασφαλίσουμε μια απόφαση η οποία θα οδηγούσε και σε λειτουργικές ε, συμπράξεις αλλά και σε μείωση του κόστους. Και έτσι η πρόταση των κρατών μελών δεν μας φάνηκε ικανοποιητική. Ε, βεβαίως όμως αν θέλετε μια γραπτή απάντηση ίσως να είναι πιο σκόπιμη. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ακούσαμε την, τις παρατηρήσεις των δυο εισηγητριών για τις εκθέσεις αυτές. Απαλλαγή λοιπόν 2012. Ακούσαμε και την Επιτροπή. Έξι εκθέσεις. Η κυρία Γκόντς. Πρόεδρε, δύο λόγια μόνο και όδηση για την απαλλαγή και εκ μέρους ομάδας μου. ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις εκθέσεις, θα καταθέσουμε στους κάποιες τροπολογίες, αλλά πάντως είναι καταρχήν ε, θετική αξιολόγησή μας. Για τη μεταφορά της έδρας της ΣΥΠΟΛ και τα όσα αναφέρονται στην έκθεση Για να είμαστε και συνεπεί στην απαλλαγή, νομίζω ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε κάποιες παρατηρήσεις για το 2012. και την ανάγκη για συγχώνευση και μεταφορά της έδρας της ΥΠΟΛ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εκφράσουμε θέσεις και για την EDPS και το πρόβλημα που την αφορά. Θα δούμε πώς θα διατυπώσουμε τις ε, ε εκθέσεις, τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ κύριε Γκόντς. Αυτά προς το παρόν. Το επόμενο θέμα στη μερική διάταξη αφορά τη συζήτηση οικονομικών ζητημάτων. Ο κύριος Δελιόγκ είναι εδώ, ο εισηγητής μας. Αλλά όχι οι άλλες δύο συνεισηγήτρες, κυρία Ρομέρο και κυρία Βέμπερ. Προτείνω λοιπόν μία σύντομη διακοπή. Μισή ωρίτσα. Μια και είχε προβλεφθεί για τις 11.30 ε, λέει ο Πρόεδρος το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Πάντως Επισημαίνω ήδη πως η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την απαλλαγή του 2012 προσδιορίζεται για τις 27, 27 Ιανουαρίου. 27 Ιανουαρίου. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Κάνω ένα διάλειμμα λοιπόν μισή ώρα. Βλέποντας ότι η κυρία Ρομέρο σκόπευε να αποχωρήσει και ότι η κυρία Βέμπερ δεν έχει έρθει, θα έλεγα ότι σκοπούμε τώρα να κάνουμε μια διακοπή για μισή ώρα και γυρνάμε στις 11.30. Be seated, please. We had done our best to mind the schedule of the order of day so that there would be a coincidence in the... Αλλάξαμε το πρόγραμμα, αλλά μαζέψαμε τους ΣΥΤΕΣ, τον κύριο Τεγιόγκ, τον κύριο Βέβερ, Περιμένουμε την κυρία Ροπέρο. Όμως, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα έρθει. Οπότε, κοινή συζήτηση των σημείων 15, 16 και 17 όσον αφορά καταρχήν το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης, ο κύριος Κορνέλης Τεγιόγκ, τεκμήριο αθότητας το 16, κυρία Ρένατε Βέμπερ και νομικές διασφαλίσεις για τα κατηγορημένα παιδιά σε ποινικέ διαδικασίες. Κυρία Κάρμεν Ρομέρο Λόπεθ. Το πακέτο το παρουσίασε η Κομισιόν πρόσφατα τονίζοντας τα δικονομικά δικαιώματα κατηγορουμένων σε ποινικέ διαδικασίες. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τον χάρτη πορείας που ξεκίνησε το 2009 με τον οποίο θεσπίζονται κοινά πρότυπα για δίκαιη δίκη. Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, τον δρόμο για την ολοκλήρωση του χώρου ελευθερίας και δικαιοσύνης. Θα συζητήσουμε τρεις πτυχές των δικονομικών δικαιωμάτων. Καταρχήν, θα ακούσουμε τον κύριο Ολιβιέ Τέλ από την Ινική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και μετά θα δώσουμε το λόγο στους συζητητές. Η Κομισιόν παρακαλώ έχει το λόγο. Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστώ τη ΛΥΜΠΕ για την διοργάνωση της σχετικής συζήτησης. Εκφράζω την ικανοποίησή μου επίση για τον λυσμό τριών εισηγητών για τις τρεις προτάσεις οδηγίας. Όπως προείπατε, Πρόεδρε, η Κομισιόν έλαβε πολιτική εντολή να φροντίσει για τα δικονομικά δικαιώματα για την εξασφάλιση δίκαιης δίκης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια βήμα προς βήμα διαδικασία. Ήδη τρεις οδηγίες εκπονήθηκαν εν προκειμένου όσον αφορά την διερμηνία, τη μετάφραση, Είναι μια οδηγία που ισχύει τον Οκτώβριο του 2013. Μια άλλη αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης για το κόστος θα ισχύσει από τον Ιούνιο και βέβαια το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο και επανένωση με την οικογένεια ή τρίτους των κατηγορουμένων και που θα υλοποιηθεί θα σωματωθεί από τα κρατημέλη πριν από τον Νοέμβριο του 2016. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 2013 για να ενισχύσει περαιτέρω τα σχετικά δικαιώματα παρουσίασε νομοθετική δέσμη μέτρων τριών οδηγιών με τις οποίες ενισχύονται εν το τεκμήριο της αθότητας. Για παράδειγμα, και με, ναι, παραδείγματος χάρη να εγγυηθεί το δικαίωμα παράσταση στη δίκη, μία οδηγία για ειδικέ εγγυήσεις για τα παιδιά, όταν είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι και μία ε, οδηγία για τα άτομα που στερούνται την ελευθερία τους και που θα πρέπει να λαμβάνουν ε, νομική αρρωγή ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Σύλληψης. Θα πρέπει η δράση της Ένωσης να είναι αναλογική. Ε, εκδώσαμε και δύο συστάσεις για τα δικονομικά δικαιώματα των ευπαθών ατόμων και μία σύσταση για την νομική αρρωγή με σκοπό να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ των εθνικών συστημάτων ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της νομικής αρρωγής. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα περάσω πάρα αυτά στην παρουσίαση των τριών οδηγιών. Καταρχάς η οδηγία για το τεκμήριο της αθωότητας. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι το θεμέλιο όλου του ποινικού συστήματος και η πρόταση είναι το θεμέλιο των δικονομικών δικαιωμάτων που υπάρχουν ήδη στην οδηγία. Η πρόταση λοιπόν για το τεκμήριο θότα έχει στενή σχέση με την ισχύουσα οδηγία και με τις δύο άλλες οδηγίες που πρότεινε η Κομισιόν για τα Δικαιώματα των Παιδιών και την Νομική Αρρωγή. Αυτές οι πτυχές είναι άρρηκτα δεμένες και είναι απαραίτητο να ανεπτύξουμε τα δικονομικά δικαιώματα ώστε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαία αναγνώριση. Η πρόταση βασίζεται στην νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όταν κρίναμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ελάχιστους κοινού κανόνες για να εξασφαλίσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη, κάναμε αυτές τις προτάσεις. Αυτή η πρόταση για την, το τεκμήριο της αθωότητας ε, θα ενισχύσει τα δικονομικά δικαιώματα που υπάρχουν στις οδηγίες. Ειδικά το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Αυτή η πρόταση έχει μία πτυχή που δεν αφορά 100% τεκμήριο της αθεότητας, αλλά είναι σημαντικό για μια δίκαιη δίκη το δικαίωμα να παρίσταται κανείς στην δίκη του. Το επίπεδο εγγύσεων στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το τεκμήριο της αθωότητας γενικά είναι υψηλό, αρκετά αποδεκτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σημεία αδύναμα όπου θα πρέπει να ισχυθεί η προστασία και διαπιστώσαμε ότι παρά τις νομοθεσίες που υπάρχουν γίνονται πολυάριθμες παραβιάσεις του, ε, του τεκμηρίου της, αθ, της στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση στηρίζεται σε τέσσερα στοιχεία. Πρώτο στοιχείο. Με βάση την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν πρέπει να επιτρέπουμε δημόσιες ακροάσεις, δηλαδή μια διοικητική αρχή ή η αστυνομία, ας πούμε, δεν μπορεί να επιτρέπει την καταδίκη ενός ανθρώπου πριν καταδικαστεί αυτός οριστικά. Θα πρέπει να προβλέπουμε δηλαδή την προστασία της φήμης του κατηγορούμενου. Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχύσουμε την βασική αρχή του ποινικού δικαίου που είναι ότι το βάρος της απόδειξης βαραίνει αυτόν που κατηγορεί και όχι αυτόν που κατηγορείται, όχι την υπεράσπιση. Υπάρχουν όμως κάποιες εξαιρέσεις. Η διαφορά ποια είναι ότι πέρα από την οδηγία που βεβαίω αντικατοπτρίζει τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πιστεύουμε ότι με την πρότασή μα θα εξασφαλίσουμε και το σεβασμό τη δίκαιη δίκη. Καλύτερο σεβασμό, εν πάση περιπτώσει, σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό που υπάρχει στην καρδιά αυτή τη πρόταση και είναι το πιο σημαντικό θέμα είναι το δικαίωμα σιωπή. Το δικαίωμα να τηρήσει κανεί σιγή όταν κατηγορείται, το να μην το να μην αυτοκατηγορηθεί και να μην ε, συνεργαστεί με την κατηγορούσα αρχή είναι βασικά, βασικές αρχές ε, για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη δίκη. Η οδηγία θα εξασφαλίσει ότι οι ύποπτοι κατηγορούμενοι δεν μπορούν να εξαναγκαστούν να προσκομίσουν αποδείξεις, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταδίκη, άδικη ή σε ε, λάθη της δικαιοσύνης. Η οδηγία όχι μόνο σέβεται αυτές τις αρχές, τις καταξιώνει, αλλά προβλέπει και κύρωση σε περίπτωση που υπάρχει παράβαση της αρχής της διατήρησης της υγιής. Όλες οι αποδείξεις ε, που λαμβάνονται ε, κατά παράβαση αυτών των δικαιωμάτων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να στηρίξουν μια καταδίκη. Τελευταίο στοιχείο αυτή τη ε, οδηγία είναι το δικαίωμα να παρίσταται κανεί στη δίκη του. Η οδηγία μιλά για μια βασική αρχή του δικαίου, τη χρησιμοποιεί και υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί, ούτω ώστε η δικαιοσύνη να μην καθυστερεί αδίκως από κακόπιστους. Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση αυτού του δικαίου, υπάρχει κύρωση, ε, υπάρχει δικαίωμα επανάληψη τη δίκη. Πάω τώρα στην οδηγία για τα παιδιά. Όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα διεθνή, αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά είναι ευπαθή άτομα λόγω τη μικρή του ηλικία και λόγω του ότι έχουν άλλη φυσικά προσωπικότητα, η οποία δεν είναι ακόμη πλήρη, είναι ατελή. Υπάρχει μια πολιτική συνένεση για την ανάγκη να προστατεύσουμε περισσότερο του ανήλικου στι ποινικέ διαδικασίε. Οι τρει ισχύουσε διαδικασίε καλύπτουν ήδη τα δικαιώματα των ανηλίκων, αλλά δεν αρκούν όμω. Δεν είναι απόλυτα επαρκή για να εξασφαλίσουμε την ειδική προστασία που χρειάζονται και να λάβουμε υπόψη τι ανάγκε που έχουν τα παιδιά σε ποινικέ διαδικασίε. Γι' αυτό ακριβώ κάνουμε αυτή την πρόταση οδηγία παράλληλα με μία σύσταση με σκοπό να προστατεύσουμε τα ευπαθή άτομα. Η οδηγία για τα παιδιά θέλει να θεσπίσει ελάχιστους κανόνες για όλα τα παιδιά, τα άτομα που είναι κάτω των 18 χρονών, τα οποία είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για, μια, για ένα δίκημα. Θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους με τρόπο κατανοητό σε αυτά, οι γονείς τους θα πρέπει να τα ενημερώσουν. Ε, τα παιδιά δεν θα πρέπει να παρετούνται από το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, γιατί δεν καταλαβαίνουν τη σημασία των πράξεών τους και προβλέπουμε ε, ένα σημαντικό το μηχανισμό, το πιο σημαντικό μηχανισμό, την υποχρεωτική υπεράσπιση από δικηγόρο για τους ανηλίκους που είναι ύποπτοι κατηγορούνται. Προβλέπεται μια κατά περίπτωση ε, αξιολόγηση της προσωπικής και οικογενειακής τους κατάστασης πριν από την ε, δίκη, ούτως ώστε να προσαρμόσουμε το, την ποινή στο αδίκημα αλλά και στην προσωπικότητα. Θα πρέπει να εξεταστούν από γιατρό αν υπάρχει ποινή δική της ελευθερίας τους και θα πρέπει να τα ανακρίνει η αστυνομία με τρόπο πολύ ειδικό. Ε, προβλέπουμε ε, οπτικοακουστική ανάκριση από την αστυνομία. Οι δικαστικές αρχές οι οποίες ε, εξετάζουν παιδιά θα πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση, θα πρέπει να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή των ανηλίκων και θα πρέπει να διευκολύνουν την επανάταξή του στην κοινωνία. Και τέλο, και σημαντικό, για το Κοινοβούλιο, οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν και εναλλακτικά μέτρα, ως προς, όχι μόνο φυλακή δηλαδή, και φυλακή μόνο κατά εξαίρεση. Όταν κρατείται ένας ανήλικο, θα πρέπει να προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως ούτω ώστε να τον εξασφαλίσουμε, να εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητά του και ζητούμε οι ανήλικοι να διαχωρίζονται πάντα από τους ε, ενήλικους ε, όταν κρατούνται. Ε, έτσι δημιουργείται και η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τα δικαιώματα των παιδιών. Σε ό,τι αφορά την τελευταία οδηγία για το δικαίωμα προσφυγής στην νομική αρρωγή, η οποία, συνδέεται άρρηκτα βέβαια με την πρόσβαση στο δικηγόρο. Υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο και προβλέπει, η τελευταία, για την πρόσβαση σε δικηγόρο υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο. Αν τα άτομα αυτά ε, στερούνται τη ελευθερία του, δεν έχουν πόρους, το δικαίωμα πρόσβασης ε, στο δικηγόρο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Εκτός και αν το κράτος δώσει εγγυήσει ότι υπάρχει αυτή η νομική αρρωγή και αυτός είναι ο στόχος της οδηγίας. Πάντα εδώ θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αρχή της αναλογικότητας. Γι' αυτό η οδηγία έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογή σε άτομα τα οποία κρατούνται, γιατί σε αυτή την κατάσταση ύποπτη είναι σε πιο, στην πιο ευάλωτη θέση και θεωρούμε ότι όταν κρατούνται η πρόσβαση σε δικηγόρο είναι ζωτική σημασία για να προστατεύσουμε την δίκαιη δίκη και κυρίως το δικαίωμα στο να μην υπάρξει αυτοκατηγορία. Τα άτομα στα κρατητήρια δεν θα πρέπει να περιμένουν για να δουν δικηγόρο και θα πρέπει οι αρχές να ορίσουν δικηγόρο. Η οδηγία προβλέπει λοιπόν μια άμεση προσωρινή νομική αρρωγή, δηλαδή δικηγόρο αμέσως. Δεν μπορούμε να ανακρίνουμε ένα άτομο όσο αυτός δεν έχει δικηγόρο που να τον έχει υποδείξει το κράτος. Φυσικά το κράτος εν συνεχεία μπορεί να καλύψει το κόστος αυτού του δικηγόρου, εάν ε, εν συνεχεία ο κατηγορούμενος αυτός δεν έχει ε, πόρους. Όλα αυτά αφορούν άτομα τα οποία αποτελούν αντικείμενο α, ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούμε όλα αυτά τα άτομα, υπόπτους και κατηγορούμενους που υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που στερούνται της ελευθερίας τους, χωρί... υπάρχει το δικαίωμα να μην αυτοκατηγορηθούν, να παραμείνουν ε, σιωπηλοί, καθώς και όλα τα δικαιώματα που αφορούν την ποινική δίκη. Επίσης υπάρχει και μια σύσταση, η οποία σκοπό έχει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σύγκληση των ε, εθνικών δικαστικών συστημάτων νομική αρρωγή, που είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ του, πολύ περίπλοκα. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι σε μια πρώτη φάση είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή τη σύσταση. Αυτέ οι δύο συστάσει μαζί θα αξιολογηθούν και αν χρειαστεί η Κομισιόν θα κάνει νομοθετικέ προτάσει για το πεδίο εφαρμογή ε, των συστάσεων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή και τώρα παρακαλώ τους οι συγητέ, τις εισηγητρίες, τους να ξεκινήσουν. Ο κύριος Κορνάλης καταρχά, καταρχάς, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που έχω να λάβει την εισήγηση για το θέμα, που είναι πολύ σημαντικό, όπως άλλωστε και η Επιτροπή κατέστησε σαφές Εάν δεν προσφερθεί ε, η δικαστική αρρωγή όπως προβλέπεται, δεν μπορούν να ασκηθούν σωστά τα ένδικα μέσα. Όλα αυτά λοιπόν είναι αρκετά περίπλοκα ζητήματα. Βρισκόμαστε προς το τέλος της θητείας. Υπάρχουν κρατημέλη τα οποία μας λένε ότι οποιαδήποτε πρόταση έχει υποβληθεί έχει επιφέρει σημαντικό κόστος. Η Επιτροπή επίσης επαναλαμβάνει ότι σε περίοδο εξυγίανσης των δημοσιονομικών είναι δύσκολο αυτό. Άλλωστε και στις κάτω χώρες ακόμη η δικαστική αρρωγή έχει τόσο πολύ απογυμνωθεί από την ουσία της που δεν μπορούμε πια να μιλάμε για δίκαιη δίκη. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και σε άλλες χώρες βέβαια. Είναι μια δύσκολη φάση όπως είπα της ε, νομοθετικής διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε με πολύ μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα. Εγώ θα περίμενα να δοθεί ιδιαίτερη ε, προτίμηση σε μια κάποια διάχυση των θεμάτων και κατακαιρματισμό τους. Εγώ όμως προτιμώ να γίνει μία ενιαία προσέγγιση και μία μόνο πρόταση. Τώρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες προτάσεις εκθέσεων. Για τη δικαστική συνδρομή, για τη νομική συνδρομή ε, είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τους νομικούς σε ποιο βαθμό μπορεί να αξιοποιηθεί το σύστημα αυτό στο πλαίσιο της οδηγίας. Η Επιτροπή βεβαίως μας λέει ότι είναι πολύ ευαίσθητα τα θέματα αυτά για τα κράτη-μέλη. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και διερωτώ με εάν τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν την ε, προσφορά των υπηρεσιών αυτών από δικηγόρους. Φυσικά υπάρχουν και ποιοτικά κριτήρια για την παροχή της ε, συνδρομής. πέραν του δικαιώματο. Βεβαίω υπάρχει και η ποιότητα τη πρόσβαση στην ε, νομική συνδρομή. Δεν αναφέρεται σαφώ στην οδηγία το τι μέσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. γιατί ανάλογα με την ε, περίπτωση μπορεί ένα κράτος μέλος να προσφέρει την νομική συντροφή ενώ σε κάποιο άλλο να μην ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι λοιπόν πολύ άνηση η εικόνα που βλέπουμε στα κράτη-μέλη και χρειάζεται να διευκρινίσουμε περισσότερο την κατάσταση και θα ήθελα πλέον πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Γιατί πάλι είναι πολύ ευρύ το πεδίο. Εγώ θα ήθελα και στο κράτος ε, της αίτηση και στο προσώοι αίτηση να υπάρχει ένας ε, συνδυασμός και μια εξίσωση των καταστάσεων. Αυτά νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες άτυπες συζητήσεις για συνεννόηση και συντονισμό των προσπαθειών με τους και ηγητές, αλλά πάντως χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις από την Επιτροπή. Και βέβαια πρέπει να δούμε τι φρονεί το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας, ε, οι πολιτικές ομάδες, για την προσέγγιση που θα επιλέξουμε. Θα προτείνουμε σύσταση για την οδηγία, πώς θα το ενσωματώσουμε στην έκθεση. Και βέβαια θέλω να δω πόσες πολιτικές ομάδες ακόμη σκοπεύουν να λάβουν το λόγο, να τοποθετηθούν στο θέμα αυτό. Δεν τρέφω ψευδεστήσει. Δεν πιστεύω ότι μέχρι το τέλο τη αιτία θα έχουμε μπορέσει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο, αλλά ίσω μπορούμε να οργανώσουμε πιο εντατικέ συναντήσει και συνεννόηση με του σκιώδει ηγητέ και να δούμε πώ μπορούμε να οργανώσουμε αυτό το κείμενο ψηφίσματο για την Ολομέλεια τουλάχιστον. Αν μπορέσουμε να πάμε και πιο πέρα, μακάρι. Εγώ είμαι στη θέσή σα για το θέμα αυτό, να εργαστώ όσο χρειάζεται, αλλά ίσω θα είναι δύσκολο να προσδοριστεί η θέση του Κοινοβουλίου για, από την Ολομέλεια, δεδομένου ότι είναι τόσο περίπλοκο όλα τα θέματα. Πάντως είμαι στη διάθεσή σας για να αφιερώσω όλο μου το χρόνο στις επόμενες εβδομάδες και να προχωρήσουμε ή δυνατόν στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος δεν ακούγεται. Η κυρία Βέμπερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε να κάνουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων για το σύνολο αυτών των μέτρων. Θα ήθελα ξεκινώντα να πω ότι είναι πολύ ωραίε πάντα οι αρχέ και απαραίτητε. Αλλά πιο πολύ εμένα με απασχολούν οι εξαιρέσει από του κανόνε. Καθώ ο διάβολο πάντα κρύβεται στι λεπτομέρειε. Και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη αυτή ανακοίνωση Υπάρχουν εδώ πράγματα τα οποία προφανώς ε, αντιβαίνουν στο στόχο των ίδιων, στη στόχευση της οδηγίας. Η Επιτροπή επικεντρώθηκε μόνο στα θετικά, τις αρχές. Εγώ πάλι, επί τη ευκαιρία, θα υπογραμμίσω ένα-δύο θέματα που μου φαίνονται πολύ προβλησιαυτοί. Υπάρχουν και περισσότερα, ομολογώ, απλώς κάποια βλέπω να φαίνονται για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφού δηλώθηκε λοιπόν ότι το βάρος απόδειξης το φέρει η διώκουσα αρχή, έρχεται ένα πλην Και το πλην λέει ότι δεν θα πρέπει η αντιστροφή του βάρους απόδειξης να είναι ε, να αποβαίνει εις βάρος της στήρησης του τεκμηρίου της αθωότητας. Με εντυπωσιάζει πολύ αυτό και αθώς στηρίζεται όλος αυτός ο συλλογισμός σε ένα και μόνο σε μια και μόνο απόφαση του δικαστηρίου του 1988 παρακαλώ ε, και μάλιστα δεν είναι καν, ε, δεν είναι καν ακριβής η αναφορά στην υπόθεση Αλαβάκου κατά Γαλλίας, γιατί πάλι ε, λέγεται ότι κάποιες υποθέσεις δεν είναι συμβατές με τον στόχο του άρθρου 6. Βλέπω λοιπόν σοβαρά προβλήματα στην υπόθεση αυτή και επίσης υπάρχει και άλλη γνωμοδότηση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, όπου πάλι μας λέει ότι είναι πολύ προβληματικό το να ανατρέπεται το βάρος της, να αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις που μάλιστα σε υποθέσεις που αφορούν ε, ανηλίκους, ε, όπου τα πράγματα ασφαλώς είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι όταν πρόκειται για ενηλίκους. το άλλο πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι στην παράγραφο 17 εκεί όπου λέγεται ότι αδίποτε προσπάθεια να υποχρεωθεί ο κατηγορούμενος ή ύποπτος να προσφέρει στοιχεία, δηλαδή, δηλαδή η υποχρέωση επιτρέπεται αλλά δεν θα πρέπει να ε, πέραν του. Αυτό είναι καινούριο. Τώρα, εάν θέλετε να εισάγουμε το Patriot Act όπως έχει, copy-paste, να το συζητήσουμε με διαφορετικούς όρους. Στη δική μου χώρα πάντως και την νομοθεσία μας η... και φαντάζομαι και στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών δεν επιτρέπεται ο εξαναγκασμός σε αυτοενοχοποίηση. Συνεχίζει η Επιτροπή όμως και μιλάει και για την αρχή της αναλογικότητας, την ανάγκη του εξαναγκασμού προκειμένου να εξασφαλιστούν στοιχεία αποδεικτικά για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος κτλ. Κοιτάξτε, εγώ έχω εργαστεί για 30 χρόνια ως δικηγόρος ε, υπεράσπιστης, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχω δει ακόμα και να παίρνουν από μια οικογένεια τα παιδιά του κατηγορουμένου προκειμένου να τον εξαναγκάσουν να δώσει στοιχεία. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση λοιπόν της Επιτροπής είναι ασαφής, επικίνδυνη υπό τις συνθήκες αυτές γιατί μπορεί να προξενήσει, να γεννήσει καταστάσεις απαράδεκτες και θα πρότεινα μετεπιτάσεως, πριν προχωρήσουμε περαιτέρω στην υπόθεση αυτή, να ετοιμάσουμε μια γνωμοδότηση, να κοιτάξουμε, να ζητήσουμε μια γνωμοδότηση τη ε, Υπηρεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πόσο είναι συμβατό με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βέβαια, βέβαια την ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή συζητεί την προσχώρησή της στην ε, Συμφωνία την Ευρωπαϊκή, των Ανθρωπινών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άρα το, το ΕΔΑΔ ε, και την υπαγωγή στη δική του νομολογία. Βεβαίως, νομικέ πτυχές πρέπει να τις συζητήσουμε και μετά, πολύ ευχαρίστω, να ζητήσουμε και μια μελέτη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για το ίδιο θέμα από επιστήμονες. Στα όσα είπε ο κύριος Δε Ιόγκ και τη δυνατότητα να εργαστούμε με ένα χρονοδιάγραμμα Ίσως ε, μπορούμε βέβαια να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο εργασίας πριν το τέλος θητείας, αλλά η ουσία της δουλειάς ε, ε, στο έργο αυτό ασφαλώς θα αφορά το προσεχές κοινοβούλιο. Αλλά υπάρχει πολλή δουλειά ούτως ή άλλως. Καλώς. Κύριε Ρομέρο, παιδιά, κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ. Και εγώ λυπάμαι που η Κομισιόν μας παρουσίασε αυτή την πρόταση για τις δικονομικές εγγύσεις. Την παρουσίασε πολύ αργά, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Θα μείνουμε στη μέση. Ήδη έχουμε προχωρήσει με τον οδικό χάρτη. Ε, κάποια θέματα εκεί υπήρχαν, ήταν αρκετά επίμαχα. Ε, τώρα με αυτές τις προτάσεις βλέπουμε τα ίδια επίμαχα θέματα να ξαναεμφανίζονται που αφορούν τώρα τις οικονομικές εγγύησεις, τους ανήλικους, την προσφυγή σε νομική αρρωγή κτλ. Εμείς πολεμήσαμε ούτω ώστε να είναι όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Γιατί δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ίσοι ενώπιον του νόμου αν δεν έχουν τα ίδια οικονομικά μέσα ή μάλλον αν λόγω διαφορετικών οικονομικών μέσων δεν έχουν τα ίδια δικονομικά δικαιώματα. Και αν δεν εποφελούνται όλοι από τις ίδιες εγγύησεις, από τα ίδια δικαιώματα κτλ. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα, ε, αυτά τα πράγματα τα οποία είχαμε ξεχάσει, τα οποία είχαμε αφήσει απ' έξω, είναι κρίμα που δεν τα ενσωματώσαμε τώρα στις δικονομικές εγγύησεις. Και μάλιστα δεν ολοκληρώσαμε τη δουλειά σε αυτή την νομοθετική, σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο για το θέμα των ανηλίκων. Πέρα από αυτά που είπε και παρά από αυτά που είπε η Κομισιόν, θέλω να πω το εξή. Υπήρχαν κάποιε εγγύησει που δεν τι είχαμε σκεφτεί καλά. Παραδείγματο χάρη την πρόσβαση στο δικηγόρο. Τα θέματα τα οποία είχαν μείνει εκκρεμή και δεν τα είχαμε σκεφτεί καλά θα μπορούσαμε να τα βάλουμε σε αυτή την οδηγία για τους α, ανήλικους. Παραδείγματο χάρη την ιατρική εξέταση. Αυτή δεν την προβλέπαμε για τους ενηλίκους, και τους ενήλικε, συγγνώμη, Επίση, τι γίνεται με την νομική βοήθεια, θα την κρατήσει κάποιο, ε, θα του την αφαιρέσουμε. Και αυτό πάλι δεν είναι σαφές. Αυτά τα θέματα τα αφήνουμε να ρυθμιστούν πότε, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Η Κομισιόν αποφάσισε αυτά που ακούσαμε. Αλλά δεν καταφέραμε το πακέτο των εγγύσεων να εμπεριέχει όλες τις εγγύσεις που θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα και μερικούς συναδέλφους που σηκώνουν το χέρι. Κυρία Ματσίου πρώτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Για να αναφερθώ σε αυτήν την πρόταση μέτρων που προτείνει η Επιτροπή, το σύνολο μέτρων που προτείνει η Επιτροπή, που έρχεται με καθυστέρηση πρέπει να πω. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές ε, δικονομικές εγγυήσεις ε, και θα έπρεπε να έχουν προταθεί ε, τα συγκεκριμένα μέτρα μαζί με το δικαίωμα της πρόσβασης σε δικηγόρο. Όπως είπε και ο κύριος Δεγιόγκ, είναι κρίμα το ότι έχουμε τέτοια καθυστέρηση. Δυστυχώς όμως με τους μισή μήνες που μας μένουν από την εντολή μας για να ολοκληρώσουμε τις προτάσεις οδηγίας και να ήμασταν, δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα θέματα τα οποία έχουν τόσο μεγάλη σημασία για το ε, λειτουργία της δικαιοσύνης. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό γιατί στην αρχή της θητείας μας είχαμε επιληφθεί διαφορών θεμάτων της λειτουργίας δικαιοσύνης και αυτό θα ολοκλήρωνε τη μεταρρύθμιση. Εν πάση περιπτώσει, το τεκμήριο της αθωότητας λοιπόν αφορά μια βασική εγγύηση, ε, αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως και εγγύησεις για τα παιδιά, όπως και η νομική συνδρομή και λυπούμε ιδιαίτερως που δεν μπορούμε ε, να ολοκληρώσουμε τα θέματα πριν από το τέλος της θητείας μας. Βέβαια συγχαίρω και την Επιτροπή που έκανε τουλάχιστον τον κόπο να τα, να τα υποβάλει ως προτάσεις, ε, έστω και τώρα. Η κυρία Σίπλε έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω μια προκατακτική παρατήρηση καταρχάς. με σκιώδη συγγήτρια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βλέποντας με πόσο κόπο και χρονοτριβές διατυπώνεται το φύλλο πορείας για, τα, για τις οικονομικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα στην περίπτωση αυτή, οφείλω να πω ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για το θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής εισαγγελία, η οποία θα μπορέσει να αναπτύξει το δυναμικό της και την αποτελεσματικότητά της μόνο όταν έχουν διατυπωθεί οι όροι για, όλη, για όλο το φάσμα των δικαιωμάτων ώστε να ασκούνται αυτά πλήρως και να εξασφαλίζονται κάποιοι ελάχιστοι κανόνες, πράγμα το οποίο δεν βλέπω να συμβαίνει. Έχω πάντως ε, ε, την πρόθεση να κάνω κάποιες παρατηρήσεις προκειμένου να βοηθήσω στην πρόοδο, να προοδεύσει συζήτηση. Καταρχάς, το πρώτο θέμα που θα αναφέρω είναι στα δικαιώματα των παιδιών. Σε διάφορους τομεί, αλλά και στο φιλοπορία, έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν ιδιαίτερε απαιτήσει όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Και αυτά θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τα κωδικοποιήσουμε, να τα ενοποιήσουμε. Ε, από την άλλη, και πέραν αυτού, βλέπω ότι δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα για άλλε ευάλωτε ομάδε. Φερρυπίν, ε, άτομα με περιορισμένη αντίληψη πνευματική, δηλαδή ενήλικους και υγιείς, οι οποίοι όμως έχουν ε, προβλήματα αντίληψης. Αυτά λοιπόν θα έπρεπε νομίζω να τα καλύψουμε. Το τεκμήριο της ε, αθωότητας είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός, πιστεύω. Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να γίνει οδηγία στον τομέα αυτό, διότι πρόκειται για ένα κύριο εργαλείο που έχουν αξιοποιήσει τα κράτη δικαίου προκειμένου να αποτρέψουν κατά ε, στρατηγήσεις, χρήσεις εις βάρος του κατηγορουμένου. Γιατί μπορεί να μην έχω στη θέση μου όλα τα αποτεκτικά στοιχεία και ε, όλα τα στοιχεία του φακέλου και να μην σε θέση να αποδείξω ότι είμαι αθώος. Γι' αυτό πρέπει η κατηγορούσα αρχή να ε, αποδείξει ότι είμαι ένοχος και όχι εγώ ότι είμαι αθώος. Επίσης, το δικαίωμα να μην αυτοενοχοποιείται κάποιος είναι πάρα πολύ σημαντική αρχή. Δεν μπορεί κάτι που έχει πει ο κατηγορούμενος να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του. Είναι νομίζω αλληλένδετο με το τεκμήριο της αθωότητας το δικαίωμα αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να παραβιάζει αυτή την αρχή και επίσης βέβαια και το να μην ε, καταδικάζεται δημοσία κάποιος πριν έχει ακόμα αρχίσει η δίκη του. Ένας ύποπτος ή απλός κατηγορούμενος δεν θα πρέπει να κάθεται στο δημόσιο εδόλιο του κατηγορουμένου γιατί παραβιάζεται έτσι η αρχή της, ε, του τεκμηρίου της αθότητας. Για την νομική συνδρομή, ο κύριος Δε Ιόγκ είπε ότι εδώ θα έχουμε ίσως ένα σημείο τριβή όσον αφορά το κόστος της δαπάνε, Είναι κάτι πάνω στο οποίο έχουμε προσκρούσει πολλές φορές, Πρέπει να πω όμως ότι μου φαίνεται απαράδεκτο σε πολλούς τομείς στη δικαιοσύνη να έχουμε δώσει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη και όταν πρόκειται για την βασική αρχή του κράτους δικαίου ε, για την τήρηση των θεμελιωδών ελευθεριών, να κάνουμε, πώς να το πω και να μεταφραστεί σωστά, να κάνουμε ένα θέατρο σκιών, λέγοντας ότι α, δεν φτάνουν τα λεφτά και θα κοστίσει πολύ. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση με τα κράτη-μέλη, προκειμένου να εκφραστεί, να εκδηλωθεί η βούληση ότι θέλουν πράγματι να τηρηθούν οι δικονομικές εγγύησεις και για την εισαγγελία Βεβαίω ε, πρέπει να συζητήσουμε, για το ένταλμα, συγγνώμη, το ευρωπαϊκό πρέπει να συζητήσουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Ιόγκ, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα της συνδρομής από δικηγόρο και στο κράτος προελεύσεως, αλλά και στο κράτος το οποίο εκτελείται το ένταλμα, όπως είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε πριν από τη θητεία. Πρέπει να αρχίσουμε πάντως να συζητούμε τα θέματα και μετά τις ε, εκλογές έστω να αρχίσουμε ως κοινοβούλιο να τοποθετούμαστε ξεκάθαρα και να ζητούμε και από τα κρατη να αναπτύξουν τις θέσεις τους προκειμένου να ολοκληρωθεί το θέμα αυτής της οδηγίας. Γιατί είναι υποχρεωμένα τα κρατη επιτέλους να θέσουν σε εφαρμογή το φύλλο πορείας όπως έχει διατυπωθεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπλ και η κυρία Λάτφορντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Περί του τεκμηρίου αθόρυτος. Δύο ερωτήσει. Πεδίο εφαρμογή. Το προτινόμενο πεδίο εφαρμογή είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ύποπτα ή κατηγορούνται σε ποινικέ διαδικασίε έως την καταλήξη τους. Όμως, στα λαδικονομικά δικαιώματα βάσει του χαρτί πορείας. Αν κατάλαβα καλά τον εισηγητή, δεν ξέρω τι ισχύει. Ισχύει αυτό που κάνουμε και στις άλλες δύο οδηγίες. Λέει λοιπόν ότι ισχύει για πρόσωπα από τη στιγμή της ενημέρωσής τους ότι είναι ύποπτα ή κατηγορημένα πρόσωπα για την τέλεση αξιοποιημένων αδικημάτων κλπ. Στην πρόταση λοιπόν δεν διευκρινίζεται αυτό. Από τη στιγμή δηλαδή της ενημέρωσης, από τη στιγμή που πληροφορούνται ότι κλπ. κλπ. Ότι είναι δηλαδή οι υποπτοί ή κατηγορούμενοι. Θα ήθελα να διευκρινιστεί αυτό παρακαλώ από την Κομισιόν. Τι ισχύει εν τέλει. Γιατί ε, δεν συνάδουν οι τρεις οδηγίες εμπροκειμένου. Και στα άρθρα 6 και 7 υπηρετισμοί, κλπ. Θα ήθελα και εδώ να, να μάθω τι πιστεύει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα εκτιμώντας στο 17 και 19, στα σημεία 17 και 19 του προημίου. Στο 17 συγκεκριμένα το οποίο ανέφερε η κυρία Βέμπερ. Διαβάζω. Υπάρχουν περιοριστικά μέτρα επιβολής με σκοπό την εξασφάλιση πληροφοριών. Και αυτό σχετίζεται με το 6 και το 7 άρθρα. Μια αυτονοχοποίηση, δικαίωμα να παραμείνει κλπ. Στη μία περίπτωση λοιπόν η προσέγγιση είναι προαιρετική, στην άλλη είναι υποχρεωτική. Και κάποιες ε, μαρτυρίες λοιπόν θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές λόγω ακριβώς άσκησης βίας. Τι γίνεται μεταξύ προημίου λοιπόν και διατακτικού. Στο προημίο, στο σημείο 19, διαβάζω και πάλι το δικαίωμα της ΙΟΠΗΣ. Είναι για τον σκοπό της μη αυτονοχοποίησης. Και όμως, λίγο παρακάτω, αναφέρεται η δυνατότητα άσκησης πίεσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτονοχοποίηση. Λοιπόν, πώς συγκεράζονται όλα αυτά. Στην Αγγλία, τουλάχιστον και την Ουαλία, που είναι οι μόνες περιοχές που γνωρίζω, ισχύει το εξής. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για το δικαίωμα κάποιου να παραμείνει σιωπηλό. Βάσει και νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις σχετικές σειρές ε, με δικαστικό περιεχόμενο στην αγγλική τηλεόραση, αλλά η γνωστή προειδοποίηση όταν συλλαμβάνουν κάποιον με την οποία είστε όλοι εξοικειωμένη περιλαμβάνει και την προειδοποίηση ότι μπορείτε να επιβαρύνετε τη θέση σας αν δεν αναφέρετε κάτι το οποίο θα μπορούσατε ενδεχομένως αργότερα να χρησιμοποιήσετε υπέρ ημών. Οπότε, βλέπετε ότι υπάρχουν περιορισμοί και προϋποθέσεις στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. Το δικαίωμα λοιπόν της σιωπής φαίνεται ότι τροποποιείται. Με τρόπο περιέγραψα και μάλιστα που εγκρίθηκε από το δικαστήριο του Στρασβουργού. Η Κομισιόν τι λέει γι' αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Βέμπερ που λέει ότι χρειάζεται κάποιο σχόλιο κάποια διευκρίνηση από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το τι ισχύει. Για το κατά πόσον αυτά είναι σύμβατα με τη σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αν είναι κάτι που υπερβαίνει τη σύμβαση. Και να δούμε και το θέμα τη ε, συνοχή. Τη ε, συμβατότητα δηλαδή του προημίου με το διατακτικό. Κύριε Αργεντινή. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. για τους υπόπτους και κατηγορουμένους και την νομική αρρωγή. Η ερώτησή μου προς την Κομισιόν είναι πώς οφείλω να ερμηνεύσω τον όρο στερουμένων της ελευθερίας τους. Από πότε ισχύει αυτό. Από την πρώτη μέρα σε ένα κρατητήριο. Γιατί ακόμα δεν θεωρείται κρατούμενος το λέω πρόσωπο. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να διευκρινιστεί αυτό. Τι σημαίνει ακριβώ πρόσωπο στερούμενο τη ελευθερία του. Οπότε μετράει η στέρηση τη ελευθερία, Από ποια στιγμή θεωρείται ότι υπάρχει η στέρηση ελευθερία. Κατά τα άλλα η οδηγία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Όμω οι συστάσει πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά τη νομική αρρωγή, τη νομική συνδρομή. για την νομική συνδρομή χρειαζόμαστε μια ενιαία γενική προσέγγιση και να μην διαφοροποιείται η προσωρινή συνδρομή. Τώρα για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης η οδηγία σύμφωνα με την οποία δίνεται το δικαίωμα εξασφάλιση δικηγόρου κλπ. Θυμίζω ότι είναι δικαίωμα στο οποίο είχε αντιτεθεί η κυβέρνησή μου. Να δηλώσουμε λοιπόν εδώ, απερίφραστα, σαφώς, ότι το δικαίωμα δικηγόρου ισχύει και στη χώρα υποδοχής, στην περίπτωση έκδοσης. Πρέπει λοιπόν και στις δύο πλευρές και στις δύο χώρες, αν θέλετε, το δικαίωμα αυτό ισχύει. Το διευκρινίζω αυτό μετά από τα όσα είπε η κυρία Λάτφορτ για το Ευρωπαϊκό Ντέλμα Σύλληψης. Πρόεδρε, Κύρκοπ, να πω καταρχάς ότι πρέπει να συγχαρούμε την Κομισιόν για την πρόοδο που σημειώθηκε. το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Όλοι εδώ συμφωνούμε, θεωρώ, με την γενικότερη προσέγγιση όσον αφορά τους κατηγορουμένους ε, ποινικές διαδικασίες. Έχω άμεση πείρα του θέματος και θεωρώ ότι η πρόοδος που σημειώθηκε ε, όσον αφορά το δικαίωμα σε διερμηνία, για παράδειγμα, το δικαίωμα πλήρους ενημέρωσης του κατηγορουμένου και ούτω καθεξής, καθώς και η πρόσβαση σε δικηγόρο. Όλα αυτά είναι ζητήματα στα οποία σημειώθηκε ταχύτητη πρόοδος. Όμως ο χρόνος πιέζει, έχουμε καθυστερήσει και θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε σάρκα και ωστά στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης πριν το τέλος της θητείας μας. Συνεπώς, τα τρία νομοθετήματα που συζητούμε εδώ. Α, και εδώ η κυρία Μακεντάιρ ε, πρέπει να απασχολείται με τα παιδιά, ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ως προς τα τρία λοιπόν νομοθετήματα, το θέμα είναι το εξή. Καταρχήν για το τεκμήριο δεν υπάρχει μια αμφισβήτηση θεωρώ. Αν και φαίνεται αυτό το τεκμήριο σε ορισμένε περιπτώσει ε, να υπονομεύεται έστω και διαδικαστικό ή και επί σε ορισμένε περιπτώσει σε ορισμένε χώρε. Κύριε Λάτφορντ, αναφέρθηκε στη γνωστή δήλωση του συλλαμβάνοντος αστυνομικού για παράδειγμα προς τον ε, συλλαμβανόμενο. Ναι, βεβαίω το δικαίωμα της ε, σιωπής υφίσταται και φυσικά δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης. Σωστά όμως ε, υπόθηκε ότι αν ο κατηγορούμενος επιλέξει να μην μιλήσει, να παραμείνει σιωπηλός, και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συναγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Θέλω να πω ότι είναι μια λεπτή διαχωριστική γραμμή αφορά βεβαίω την αστυνομία και όλα αυτά θα τα λάβει υπόψη η αστυνομία. Πάντω, εν γέννη, πιστεύω ότι είναι σωστό. Οποιοδήποτε να μπορεί να παραμείνει σιωπηλό και να μην πει κάτι το οποίο θα τον ενοχοποιήσει, που θα ενοχοποιήσει ή άλλον. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αναφερθεί στο ζήτημα, το ίδιο έκανε και η Λάτφορντ. Λέω λοιπόν ότι όπως και προείπα, πρέπει να υπάρχουν ε, συναφείς εγγύησεις και υπάρχουν. ελάχιστοι πάντως κανόνες όσον αφορά τον χειρισμό των ε, υπόπτων και κατηγορουμένων ισχύουν αλλά πρέπει να τους ενισχύσουμε περαιτέρω. Χρειαζόμαστε κάποια ελάχιστα κοινά πρότυπα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πρόσβαση σε δίκαιη δίκη. Νομική συνδρομή, εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, πιο πολύπλοκα. Μετά, αλλά ξέρετε, συμφώνησα, δεν είχα ποτέ αντίρρηση, όμως με την νομική συνδρομή τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Διότι το θέμα, πιστεύω, είναι, πρέπει να είναι αντικείμενο ρυθμίσει από τα κράτη-μέλη. Γιατί ο τρόπος χρηματοδότησης διαφέρει. Κάπου υπάρχει χρηματοδότηση, κάπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα λέω ότι επηρεάζονται τα δικαιώματα του καθού κάθε φορά που, μάλλον από χώρα σε χώρα, γιατί σε μια χώρα μπορεί να μην υπάρχει υπαρκής χρηματοδότηση. Και για να κλείσω, πρόεδρε, ως προς το ευρωπαϊκό ένταμα, ένταλμα σύλληψης που όλοι λέμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί. Mm. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ναι, λέμε, ωραία να υπάρχει παντού, επαρκή νομική συνδρομή. Όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να φροντίσουμε να γίνουν σεβαστά όλα τα δικαιώματα του κατηγορμένου. Και αυτή η διαδικασία πρέπει να τροποποιείται κατά περίπτωση στην συναρτήση των αναγκών χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα ανά την Ευρώπη εργαλεία. Και σίγουρα το ευρωπαϊκό Ανταλημά σύλληψης είναι πολύ σημαντικός τομέας, μια πολύ σημαντική έννοια και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε προκειμένου να θεσπίσουμε οριζόντια μέτρα. Κύριε Μακεντάε, όσον αφορά τι αντικονομικέ εγγύσει για τα παιδιά. Και πάλι, συνιστάται προσοχή όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη νομική συνδρομή, όμω εδώ έχει ζωτική σημασία. Να διευκρινίσουμε απολύτω τι είδου πληροφορίε παρέχονται στον κηδεμόνι τους γονείς του παιδιού, είτε έχετε να εμπλέκεται η ευθύνη τους. Και έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε γίνεται για τα παιδιά είναι προσαρμοσμένο στα παιδιά, στα ανάγκες των παιδιών. Η ανήλικη είναι άλλη ιστορία. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα μεταφέρουμε αυτά αυτούσια στην περίπτωση των παιδιών. Τα παιδιά είναι διαφορετικά. Δεν είναι ενήλικοι, έχουν διαφορετικές ανάγκες χρήζουν περισσότερη προστασίας σε σύγκριση με τους ενηλίκους στις περισσότερες περιπτώσεις. Προσοχή λοιπόν, ας μην κολλήσουμε ό,τι ισχύει για τους ενηλίκους στην περίπτωση των παιδιών άκρητα. Πρόεδρος, πολύ ωραία, ακούσαμε διάφορα πράγματα, διάφορες απόψεις. Προτείνω το εξή. Η διαδικασία βρίσκεται στα πρώτερη στάδια του συζήτηση. Εμείς παρακολούθησαμε προκειμένου την παρουσίαση της Κομισιόν. Θα έλεγα να μην γίνει δεύτερος γύρος με παρεμβάσεις εισηγητών, εκτός αν θέλετε να πείτε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το καλό είναι ότι είμαστε εδώ σήμερα για να ακούσουμε και θα ακούσουμε τις επεξηγήσεις της Κομισιόν μετά από τις παρεμβάσεις των μελών και των εισηγητών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο να είστε όμως πολύ σύντομοι, διότι μας απομένει ελάχιστος χρόνος μέχρι το τέλος της ε, πρωινής συνεδρίασης. Θέλουμε και τη δική σας ε, συμβολή για να κλείσουμε στην ώρα μας. Αυτά. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Είμαστε στη διάθεσή σα να έρθουμε σε επαφή με του εισηγητέ και του κοιόδη εισηγητέ για να συζητήσουμε λεπτομερώ αυτά τα κείμενα. Για το θέμα τη νομική αρρωγή. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σα σε έναν βαθμό, αλλά λάβαμε υπόψη ότι ποικίλουν πολύ τα, τα συστήματά μα, ότι είναι περίπλοκα και βεβαίω η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση μα δημιουργεί ιδιαίτερε προκλήσει. Στα κράτη-μέλη τη δημιουργεί δηλαδή. Υπάρχει διχοτομία αυτή ανάμεσα στην οδηγία και στη σύσταση και του δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες. Για το τεκμήριο της αθότητας, ευαίσθητο θέμα. Όλες οι προτάσεις ε, βασίζονται στα, στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν είναι πολύ σαφές αυτό. Μερικές φορές θέλησαμε να πάμε παραπέρα, ειδικά σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στη σιωπή. Πρέπει να συγκεράσουμε δύο ανάγκες σε ό,τι αφορά το τεκμήριο της αθότητας. Από τη μία, να εξασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη για τα θύματα και να διωχθούν οι δράστες και από την άλλη να εξασφαλίσουμε το σεβασμό των δικαιωμάτων. Ε, γι' αυτό ακριβώς σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στη σιωπή, για να απαντήσω και στα σχετικά ερωτήματα, θεωρούμε ότι δεν μπορούσαμε να συνάγουμε συμπεράσματα από τη σιωπή ενός ανθρώπου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα από τη σιωπή. Γιατί αν λαμβάναμε υπόψη τη συγκεκριμένη επίσης νομολογία, ε, θα αποδυναμώναμε την ουσία ε, το νόημα αυτού του δικαιώματος στη σιωπή. Επομένως, δεν πρέπει να δεχτούμε τις παρεκκλήσει. Αυτό για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, η διατύπωση είναι διαφορετική για το... Τον παιδ... Η διατύπωση είναι διαφορετική και εξασφαλίζει διαφορετικά πεδία εφαρμογή. Ε, μοιάζει με, την, με το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για τον την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν χρειάζεται επίσημη ε, κοινοποίηση αυτή τη στιγμή είσαστε ένοχο. αν η αρμόδια αρχή το, σας θεωρεί ένοχο, τότε, ε, συγγνώμη, ύποπτο, τότε εφαρμόζεται η σχετική οδηγία. Τελείωσε. Αυτά. Ευχαριστώ για την ε, κατανόησή σας. Φτάσαμε στο όριό μας, 12.30. Συμπερασματικά θα έλεγα οι εισηγητές να έρθουν σε επαφή με τους και ηγητές και να τους ενημερώσουν, ούτω ώστε να αποφασίσουν τι θα κάνουμε στο μέλλον. Τι μέλη γενέστε. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Πώς θα παρακολουθήσουμε την κάθε μία από αυτές τις οδηγίες. Να σας αναγγείλω τώρα κάτι. Για πρακτικούς λόγους πρέπει να σας αναγγείλω ότι δυστυχώς θα ξαναρχίσουμε στις 3 την συνδρίασή μας, αλλά όχι εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Στο 7C50 στο PHS, από τις 3 μέχρι τις 4 αυτό, σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτήν την αίθουσα. Και εν συνεχεία, από τις 4 και μετά, μέχρι το τέλος, θα είμαστε σε άλλη αίθουσα, στο PHS, στο 3C50. Sorry, ε, συγγνώμη για αυτή την αλλαγή αίθουσας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στο PHS 7C50, από τις 3 μέχρι τις 4 και από τις 4 μέχρι τις, 6, ε, μέχρι τις στο 4. Στο PHS πάλι, στο 3 c 50.